Thank Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Προχωρούμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Πρώτη έκθεση είναι η έκθεση ΕΡΤΟΚ. Κυρία Σόιντροβα, έχετε το λόγο παρακαλώ. Μισό λεπτό μάλλον, κυρία Σόιντροβα. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, βρισκόμαστε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Παρακαλώ λοιπόν να αποχωρείτε ησύχω Κύριε Σόντροβα, έχετε το λόγο.